Bonjour à tous. La Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε. Έχετε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης στη διάθεσή σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Και επομένως τα πρακτικά υιοθετούνται. Με βάση την ημερήσια διάταξη θα περάσουμε στην κοινή συζήτηση για, το Ευρωπαϊ... για τα ευρωπαϊκά ταμεία.